Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, θα ξεκινήσουμε ε, αυτήν την κοινή ακρόαση της Επιτροπής ΔΕΒΕ και της Επιτροπής Άγκρη εκ μέρους ε, του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτήν την κοινή ακρόαση με τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας και Γεωργικής Ανάπτυξης. Ε, όπως θα ξέρετε, κοινή γεωργική πολιτική ε, θα μεταρρυθμιστεί σημαντικά με το 2020. Θα, γίνει, τα λάβει χώρα μια σημαντική μεταρρύθμιση. Έχει, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προεργασίες. Η δημόσια διαβούλευση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κοινή Πολιτική οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έδωσαν έμφαση στο θέμα της πολιτικής για την ανάπτυξη μόνο σε ένα βαθμό. Την ε, συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη. Ε, λαμβάνονται υπόψη ε, οι πρόσφατες αλλαγές βεβαίως ε, στην διεθνή συγκυρία καθώς και οι αλλαγές ε, που αφορούν ε, τις γεωρικές τιμές, διαπραγματεύσεις για εμπορικά ζητήματα αλλά και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν την κλιματική αλλαγή αλλά και το CDGS Γι' αυτό λοιπόν οι επιτροπές ΔΕΒΕ και Άγκρι αποφάσισαν να οργανώσουν αυτή την κοινή ακρόαση, τη δημόσια ακρόαση σε ό,τι αφορά ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Επιτροπή ΔΕΒΕ έχει ζητήσει επίσης μια μελέτη έτσι ώστε να αποτελέσει αυτή βάση για επικοδομητικές συζητήσεις με συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις για το πώς να θα εφαρμόσουμε, θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την ε, ανάπτυξη ε, και για την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή εν ώψη της μελλοντικής μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή, είναι η στιγμή να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις έτσι ώστε η κοινή γεωργική πολιτική να λαμβάνει όντως υπόψη την πολιτική ανάπτυξη. Θα ακούσουμε σε λίγο τους εμπειρογνώμονες, περιμένουμε μονησία την ακρόαση. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό θέλω να καλωσορίσω την Γκαμπριέλα Ζωάνα, Ζωάνα πολύ ωραία, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία θα συμπροεδρεύσουμε ε, σε αυτή την ακρόαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούλογλου στο όνομα της Επιτροπής Γεωργίας και Γεωργίας Ανάπτυξης ε, του οποίου τον πρόεδρο εκπροσωπώ και είναι τιμή μου, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμά όλους τους ε, ομιλητές που δέχθηκαν να συνεισφέρουν σε αυτήν την κοινή ακρόαση, μεταξύ των οποίων βεβαίω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αυτή η κοινή ακρόαση θα μας επιτρέψει ε, να εξετάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ε, του κατά πόσο υπάρχει αντίκτυπος της κοινή λογικής πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ποιος είναι αυτός ο αντίκτυπος, πώς έχει αλλάξει με τον καιρό. Ε, Ετοιμάζουμε να ακούσουμε ενδιαφέρον επίσης ε, τις συστάσεις για τη μέλλον της κοινής πολιτικής μετά το 2020, ε, πώς δηλαδή θα πρέπει να σχεδιαστεί η κοινωνική πολιτική έτσι ώστε να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτή τη φάση αυτά που θα υποθούν σήμερα ε, μπορούν να επηρεάσουν την μεταρρύθμιση. Μια και η διαδικασία έχει ξεκινήσει σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή μα. Με την προπαρασκευή της ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για το μέλλον ε, της διατροφής και της γεωργία. Η ακρόαση χωρίζεται σε τέσσερα κομμάτια. Πρώτα, μια παρουσίαση τη μελέτη για το αντικείμενο της ακρόασης ε, με μια παρουσίαση κάποιων συγκεκριμένων παραδειγμάτων, την παραγωγή γαλάκτος στη Δυτική Αφρική, παραδείγματος χάρη, και ο αντίκτυπος της κοινής πολιτικής στο περιβάλλον, ε, το θέμα επίσης της χρήσης της γης και της κατανάλωσης κρέατος. Το δεύτερο πάνελ ε, θα εξετάσουμε την εξέλιξη της κοινής γεωργικής πολιτικής στα πλαίσια του άρθρου 208 της συνθήκης, καθώς και τα συμπεράσματα για την πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη και την νέα κοινή πολιτική. Το πρώτο, στο πρώτο πάνελ ε, θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ, ο Στέγιος Κούλογλου, και εγώ θα προεδρεύσω στο δεύτερο πάνελ. Στο κάθε πάνελ θα έχουμε δύο παρουσιάσεις, δέκα λεπτά η καθεμία, που θα, συνεχί, που θα, τις οποίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις έχουμε μια αρκετά φιλόδοξη, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την κοινή ακρόαση σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι να σεβαστούν τον χρόνο που τους έχει ε, δοθεί. Ο καθηγητής ε, αγροοικονομικών, η ε, κυρία Μαρία Μπλάνκο από τη Μαδρίτη, θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για την αντίκτυπο της κοινή γεωργικής πολιτικής της αναψώμενες χώρας. Ε, κυρία Μπλάνκο, έχετε το λόγο, παρακαλώ. ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα τη μελέτης αυτής για την αντικτύπο της ΚΑΠ 2014 και 2020 στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καταρχάς, θα ήθελα να σας δώσω το γενικότερο συγκείμενο σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ και μετά θα κοιτάξουμε το βασικό θέμα της μελέτης μας, το οποίο και είναι η εκτίμηση του αντικτύπου της τρέχουσας ΚΑΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, θα προβούμε και σε κάποιες συστάσεις για την τρέχουσα συζητήσεις για το μέλλον της ΚΑΠ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το γενικότερο πλαίσιο. Σε βάθος χρόνου διαπιστώνουμε ότι η ΚΑΠ ανασχεδιάζεται κάθε φορά όσο ανακύπτουν και νέες προκλήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές ε, οφείλονται και σε εξωτερικές επιρροές Υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες και στα γερμανικά. Πολύ ωραία. Συνεχίζω. Έλεγα λοιπόν ότι κάποιες από τις προκλήσεις αυτές έχουν να κάνουν και με εξωγενείς παράγοντες σε ό,τι αφορά και τους αναπτυξιακούς στόχους. Στόχος μας είναι να δώσουμε υποστήριξη σε Ευρωπαίους ε, αγρότες με τρόπο που να μην ε, ε, στρεβλώνει την αγορά και να μην αμειγνύεται στην αγορά. Κοιτώντα λοιπόν την, ε, τα κονδύλια ΚΑΠ σε βάθο χρόνου στο γράφημα, διαπιστώνουμε ότι κάποια στοιχεία καθιστούν την ΚΑΠ πιο συμβατή με τους στόχους τους αναπτυξιακούς. Καταρχάς, ο τερματισμός των ε, επιδοτήσεων εξαγωγών. Βλέπετε πώς αποτυπώνεται στο γράφημα. Δεύτερο θέμα, σταδιακή κατάργηση των συνδεδεμένων πληρωμών. Αποσυνδεδεμένες λοιπόν πληρωμές και ενισχύσεις και βλέπουμε ε, ότι στην τρέχουσα κάπα έχει ανατραπεί αυτή η τάση και αυτό αποτυπώνεται το γράφημα. Τέλος, η ενίσχυση των εργαλείων προκειμένου να ανταποκριθούν σε περιβαλλοντικές ανησυχίες και στον πρώτο μα και στο δεύτερο πυλώνα. Βλέπετε στο γράφημα τις γραμμέ και την αύξηση, την ενωδική πορεία με την πάροδο του χρόνου. Από διεθνή λοιπόν άποψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μεγάλο παράγοντα στις αγροτικές και αγορές και τις αγορές τροφίμων. Σήμερα οι κοντινές σχέσεις ε, με άλλες χώρες καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό εισαγωγέα τροφίμων από χώρες ΑΚΕ σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το 11% όπως βλέπετε στο γράφημα ως ποσοστό και το εμπορικό ισοζύγιο είναι πιο θετικό όσο περνάει ο καιρός. Στην δεξιά πλευρά είναι σαφές πως είναι η εξέλιξη εξαγωγών και εισαγωγών, οι εισαγωγές από χώρες και αυξάνονται όπως βλέπετε με την πάροδο του χρόνου. Τώρα να στραφούμε στον τομέα επικέντρωσης ε, της ε, έρευνας. Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στις αναπτύξεις και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιος είναι ο αντίκτυπος λοιπόν της ΚΑΠ 2014-2020 στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εξετάζουμε κυρίως τον αντίκτυπο σε θέματα επιστημιστικής ασφάλειας, περιβαλλοντικών συνεπειών και κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών. Για να απαντήσουμε λοιπόν στο ερώτημα αυτό, αναθεωρήσαμε και εξετάσαμε τις προηγούμενες μελέτες, αναλύοντας τον αντίκτυπο της ΚΑΠ. Δεν διαπιστώσαμε πολλές μελέτες να ε, επικεντρώνονται ιδιαίτερο στον αντίκτυπο της ΚΑΠ στις ανεψόμενες χώρες. Μα υπάρχουν πολλές μελέτες, θα μου πείτε. και έχετε. Επικεντρώνονται όμως σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα ή για παράδειγμα στον αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων, αν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, αν αυξάνονται η πιστητική ασφάλεια. Αλλά δεν επικεντρώνονται στον αντίκτυπο της ΚΑΠ στις οικονομίες αυτές σε σχέση και με τον αντίκτυπο άλλων πολιτικών με παρόμοια αποτελέσματα. Και ως εκ τούτου τι διαπιστώσαμε. Ότι είναι δύσκολο να απομονωθούν ε, οι συνέπειες της ΚΑΠ σε σχέση με τις συνέπειες άλλων πολιτικών. Κάτι άλλο θετικό είναι το εξής. Φαίνεται ότι υπάρχουν σιγά σιγά στοχευμένες ε, μελέτες για τον αντίκτυπο της ΚΑΠ και ένα σημαντικό θέμα ιδιαίτερος είναι η μελέτη αντικτύπου εξάντα για την ΚΑΠ 2014 και 2020 που ήδη περιλάμβανε μία μελέτη αντικτύπου για τις τρίτες χώρες. Έστω και αν δεν ήταν. τόσο εντελεχής όσο η μελέτη αντικτύπου για τον αντικτύπο στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε μπει όμως το επίκεντρο το θέμα αυτό και αυτό αποτελεί καλή ένδειξη. Ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε λοιπόν τα βασικά πορίσματα. Καταρχάς, επιστημιστική ασφάλεια. Ποιος είναι ο αντικτύπος. Σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ, διαπιστώνουμε ότι τρέχουσα ΚΑΠ δεν τροποποιεί σημαντικά την κατάσταση. Ο αντίκτυπος ε, στις διεθνείς αγορές ε, είναι μάλλον περιορισμένος. Γιατί οι τιμές των αγροτροφίμων σε ευρωπαϊκή επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζουν λίγο πολύ με τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και άρα οι αλλαγές ε, της τρέχουσας ε, ΚΑΠ για την παραγωγή και το εμπόριο και για τις τιμές είναι ίσονος σημασίας. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, οι οποίες βασικά έχουν να κάνουν με την εισαγωγή εθελούσιας ενίσχυσης ε, ΚΑΠ. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η εθελούσια υποστήριξη σε κάποιες ε, επιχειρήσεις, αγροεπιχειρήσεις, σε κάποιους συγκεκριμένους ε, τομείς που πλήττονται από, διάφορες, από παράγοντες και αυτή η εθελούσια υποστήριξη χορηγείται για να διατηρηθεί το επίπεδο παραγωγής στις περιπτώσεις αυτές. Αριστερά στο γράφημα βλέπετε ότι η εθελούσια συνδεδεμένη υποστήριξη αποτελεί 10% του προπολογισμού άμεσων ενισχύσεων σήμερα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και βλέπετε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τα κρατημέλη το 2014, οι οποίες και τροποποιήθηκαν το 2016, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Άρα τα στοιχεία αυτά ισχύουν και σήμερα. Δεξιά βλέπετε ότι καταρχάς τα πιο πολλά κράτη-μέλη εκτός από τη Γερμανία αποφάσισαν να χορηγήσουν τελούσια συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις βασικά για ζωικά προϊόντα. Ένας άλλος ε, τομέα είναι οι πρωτενούχες καλλιέργειες. Το βλέπετε αυτό στα δεξιά. Πάνω από 40% των ενισχύσεων πάει στο βόλιο κρέας και 11% στις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια βασική ανησυχία όταν εξετάζουμε τον αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και γιατί? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία από τις λίγες μελέτες και έρευνες που αναλύουν τον αντικτύπο της ΚΑΠ. Όχι ιδιαίτερος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα μέτρο σύγκριση. Μάλλον η μελέτη, η έρευνα συγκρίνει την κατάσταση με την προηγούμενη ΚΑΠ. Ας δούμε, λοιπόν, κάποια από τα πορίσματα της έρευνας. Βλέπουμε στην πρώτη στήλη την ε, αναφορά που είναι η προηγούμενη ΚΑΠ. Στη δεύτερη βλέπουμε την ΚΑΠ 2014-2020. Στην τρίτη στήλη βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά χωρίς ε, τις εθελούσιες συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις και στο τέλος χωρίς τον πράσινο προσανατολισμό, τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Γιατί, γιατί αναλύοντας τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι η εθελούση αυτή η συνδεδεμένη υποστήριξη υποστηρίζει πολύ την παραγωγή. Δηλαδή, χωρίς το πρασινισμά και χωρίς αυτές τις ενισχύσεις θα είχαμε μείωση σε κάποιους τομείς. Αλλά από μόνη της η εθελούσια συνδεδεμένη άμα υποστήριξη υποστηρίζει την παραγωγή. Έτσι αποφάσισαν τα κράτη-μέλη δεν απασχολεί αυτό ιδιαίτερα τι αναπτύσσόμενε χώρε, αλλά αυτό ισχύει και για τα πιο πολλά ζωικά προϊόντα. Γιατί βλέπουμε ότι χωρί αυτή την εθελοσία συνδεδεμένη ενίσχυση, τι θα γινόταν. Η παραγωγή των ζωικών αυτών ε, προϊόντων θα μειώνονταν. Οι τιμές όμως θα ανέβαιναν και τελικά το αντίκτυπο θα ήταν θετικός εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το εισόδημα των γεωργών και των εκτροφέων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ποιος είναι ο αντίκτυπος πραγματικά της ε, θελούσιας συνδεμένης ενισχύσης. Αυτό λοιπόν αποτελεί μία από τις βασικές ανησυχίες όταν εξετάζουμε τον αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές και στο εμπόριο. Κοιτώντας, λοιπόν τον περιβαλλοντικό αντικτύπο. Διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει και περαιτέρω βήματα με την εισαγωγή του πράσινου προσανατολισμού, αφού του πρασινίσματος και πιο πολλών ε, τέτοιων περιβαλλοντικών μέτρων στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η αύξηση του ανταγωνισμού ...δεν είναι όφηση και στην ε, γεωργική ανάπτυξη και σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά μπορεί και να έχει και άλλο αρνητικό αντικτύπο στην βιώσιμη ανάπτυξη. Και πάλι λοιπόν η βασική κριτική ασκείται για τα ζωικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφενός ε, η αύξηση των ε, ζωικών κεφαλαίων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι αυξάνονται αντίστοιχα και η ανάγκη για ζωοτροφή, η οποία με τη σειρά της προωθεί την παραγωγή ζωοτροφών σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά αυτή η αύξηση της παραγωγής μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, μπορεί να σημαίνει επιπλέον πιέσεις στους υδατινούς πόρους και το καθεξής. Άρα υπάρχουν ανησυχίες και εδώ. Υπάρχει δε ανησυχία και για την συνοχή της υποστηρίξης ΚΑΠ με τους περιβαλλοντικούς και τους κλιματικούς στόχους, κατά πόσον συνάδουν αυτά τα δύο σκέλη. Όχι μόνο εκτός αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν υποστηρίζουμε κάποιους συγκεκριμένου τομεί και η υποστήριξη των τομέων αυτών σημαίνει ότι θα υπάρξει ανετικός αντικτύπωση για το περιβάλλον, ίσως να εφαρμόζουμε τελικά περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία είναι αντίθετα ή τουλάχιστον δεν συνάδουν με τα μέτρα υποστήριξη τη παραγωγή. Αυτέ είναι οι βασικές ανησυχίε, ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε ό,τι αφορά τώρα τον κοινωνικό και δημογραφικό αντίκτυπο. Είναι πάρα πολύ περιορισμένε δυστυχώ οι έρευνες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν υπάρχουν στοχευμένες έρευνες που να εξετάζουν συγκεκριμένα και μόνο τον αντίκτυπο της ΚΑΠ. Υπάρχουν κάποιες βέβαια που διαπιστώνουν ότι αν δεν υπάρχει στραβλωτική ΚΑΠ μπορεί να έχει αυτό θετικό αντικτυπώ στο διεθνές εμπόριο σε μεγαλύτερες εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση των εξαγωγών ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την, ε, την οικονομία της υπαίθρου και το περιβάλλον και τέλος ότι τα κριτήρια ε, επιλεξιμότητας στα περιστατικά του τρέχοντος συστήματος GSP+, μπορεί να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, αποφεύγοντας ε, τις αρνητικές επιπτώσεις για τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Δεν υπάρχουν όμως επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την αποδοτικότητα του συστήματο. αυτού. Είναι καινούριο. Θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Αυτό σε ό,τι αφορά το σκέλο το κοινωνικό και το δημογραφικό. Και θα κλείσω με κάποιε συστάσει για τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Καταρχά. υπάρχει πρόοδος για την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να επιλύσουμε. Οι βασικές προκλήσεις θεωρούμε είναι οι εξή. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις μελλοντικέ μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιμη αναπτυξιακή ατζέντα, τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εγκάρσια πολιτική. Δεν μπορούμε να τα απομονώσουμε όλα αυτά σε μία και μόνο πολιτική χωρίς να έχουμε υπόψη τα μέτρα που λαμβάνουν οι άλλοι τομείς. Γιατί η διασύνδεση μεταξύ των τομέων είναι άρρηκτη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, ασφαλώς. Αν πραγματικά θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο σημείο αυτό, θα πρέπει να μπορέσουμε να προσμετρούμε τον διατομιακό αντίκτυπο των πολιτικών. Χρειάζεται μια συστημική προσέγγιση για την αξιολόγηση, την καταμέτρηση του αντίκτυπου των γεωργικών πολιτικών, προκειμένου να λεφτεί υπόψη η επίδραση και η διάδραση σε όλους τους τομείς και για να προωθηθεί πραγματικά η πολιτική και τα εργαλεία της πολιτικής τα οποία θα δρουν σε συνέργεια το ένα με το άλλο. Αυτό και σε ιστορικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Επίσης, θα χρειαστούμε συγκεκριμένους δείκτες για να αξιολογήσουμε και να παρακολουθήσουμε τη συμβολή στην επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμη ανάπτυξη στι αναπτυσσόμενε χώρε. Θα κλείσω με τους ιδιαίτερους τομεί ανησυχία, τις ιδιαίτερες ανησυχίε μας. Να θυμάστε ότι πρόκειται για μία μελέτη, μία έρευνα, η οποία προκύπτει από αναθεώρηση προηγούμενων ερευνών. Έχω εξετάσει λοιπόν πολλούς άλλους τομείς και εδώ βλέπουμε λοιπόν τι έχει ανακύψει ως πόρισμα. Έχουμε και άλλα φυσικά, έχουμε και άλλες λεπτομέρειες στην ε, έρευνα, αλλά να σας πω ποια είναι τα βασικά απορίσματα. Καταρχάς, ότι η επανεισαγωγή της αυτελούσιας συνδεδεμένης ενισχύμη στην ΚΑΠ του 2014 και 2020 είχε αντίκτυπο στρέβλωσης της αγοράς και ιστορικά και στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα ήθελα να τονίσω ότι ιδανικά αυτές οι ατελούσιες συνδεδεμένες ενισχύσεις θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνο στους πλέον αδύναμους τομείς και στις πλέον ευάλωτες περιοχές. Κάποιες περιοχές το χρειάζονται, σύμφωνοι. Είναι περιοχέ περιοχές φυσικής ε, προστασίας, χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία, έχουν κάποια πολύ ευαίσθητα κάποιε πολύ ευαίσθητε καλλιέργειε. Για όλα τα υπόλοιπα τα προϊόντα όμω θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά αν πραγματικά χρειάζονται τα εργαλεία αυτά, το συγκεκριμένο μάλλον εργαλείο. Κατά δεύτερον, συγκεκριμένα κίνητρα για κάποια εργαλεία της ΚΑΠ σε ό,τι αφορά και τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Εδώ η βασική σύσταση είναι να ληφθεί υπόψη και η επίδραση στο περιβάλλον. Όταν υποστηρίζουμε, ενισχύουμε κάποιους τομείς. Και εδώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και το ζωικό κεφάλαιο που ενισχύονται σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο σημείο ανησυχία είναι ο βαθμό αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του νέου συστήματο GSP για να προωθηθεί η επιστημιστική ασφάλεια και για να συμβάλλουμε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι δύσκολα τα κριτήρια αυτά, περίπλοκα τα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά θα πρέπει να αποτρέπουν ε, τις αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τοπικό επίπεδο. Πολύ περιπλοκό λοιπόν αυτό και προαπαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Άρα θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά πορέσματα της έρευνας. Νομίζω ότι όλοι την έχετε στη διάθεσή σας, αν έχετε ερωτήσεις, με χαρά να τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπλάνκο. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Αντάμ Διάλο είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης μικροπαραγωγών ε, γάλακτος μα στην τροφή. Επίσης θα συζητήσουμε και το θέμα της παραγωγής γάλακτος στην Δυτική Αφρική. Καλημέρα και σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε εδώ για να, φερθεί για να αναφερθώ σε αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μου. Ε, το όνομά μου είναι Ανταμά Ανταμά Ιμπραήμ Διαλό, είμαι γαλακτοπαραγωγός αλλά και μεταποιητής εδώ και 20 χρόνια. 180 χιλιόμετρα από τη Ουαγκαντούγκου βρίσκεται η εκμετάλλευσή μου και είμαι ο πρόεδρος της ε, Εθνικής Ένωσης Παραγωγών καθώς και αντιπρόεδρος της α, Διαπαγγελματικής Ένωσης όπου η κτηνοτροφία αποτελεί 80%, απασχολεί 80% των εργαζομένων. Σημαντικός αριθμός ζώων, ε, περίπου 1 9 ε, εκατομμύρια βοηθοί πολύ σημαντικός των εξαγωγών. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής ε, βοσκοτόπων. Έχουμε μια εκτατική μορφή κνοτροφίας με περιορισμένο αριθμό ζώων ανά άνθρωπο. Ε, ουσιαστικά είναι το γάλα Είναι τόσο σημαντική η παραγωγή γαλάκτος στη χώρα Από τη δεκαετία του 90 και μετά αρχίσαμε να αναπτύσσουμε μικρά γαλακτοκομεία, μονάδες δηλαδή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, κοντά στις ζώνες παραγωγής, κοινοτρόφων, έχει υπάρξει μια αξιοποίηση οικονομική σε εμπορικό, σε τοπικό επίπεδο και για τους νέους, χάρη στα και αυτό έχει επιτρέψει στις οικογένειες ε, και στις γυναίκες ε, ε, να μπορούν να καλούν χρόνο. Αυτό είναι ένα σημαντικό διακύβευμα για μας και αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει να φτάνουν στην αγορά προϊόντα φτηνά ενώ και δεν γίνεται επαρκή προσπάθεια έτσι ώστε να προωθηθούν τοπικά, δεν προστατεύει επαρκώ τα προϊόντα μας. Υπάρχει φορολόγηση 5% για το γάλα, ε, στα πλαίσια της Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ορίζουν σε μηδενικό δασμό, 0% για το γάλα, το γάλα χίδιν. Σαν στην δημιουργία των μικρών αυτών γαλατοκομείων σε αυτή την υποπεριφέρεια, και εδώ πάντως οι επενδύσεις ε, και οι πολιτικές οικονομικών ποσοστώσεων στην Ευρώπη οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής. Στην Ευρώπη, εδώ, πάνω από 2% το 2017, προθεματοποιημένη σε ό,τι φορά το γάλα σε σκόνη. Επίσης, ε, έχουμε αύξηση της τιμής ε, του βουτύρου μέσω του γάλακτος ε, του 2017. Όλα αυτά λοιπόν τελικά είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και όχι Για να πάμε τώρα λίγο πιο γρήγορα, διαπιστώνουμε ότι ε, λίτρα γάλακτος Εάν δούμε λοιπόν το, ζήτημα αυτό από πιο κοντά, το πρόβλημα είναι, είναι πολύ πιο ακριβό. Μετά από μια μελέτη που έγινε, ε, δείχνει ότι το γάλα σε σκόνη παρακάμπτοντας τους κανόνες, διότι αυτή η παραγωγή γάλατος σε σκόνη επιτρέπεται νομίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επιτρέπεται στην Αφρική. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι συκτοχύνουμε κι άλλο. Είναι κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακόμα ε, μεγαλύτερε μεταναστευτικέ ροέ. αντίσταση σε αυτό το ρεύμα. Θέλουμε καταρχήν να δημιουργήσουμε μία μάρκα, ένα λόγο ε, που θα διαχωρίζει το τοπικό γένος δικτύου τοπικού γάλακτος ε, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιφέρεια. Και αυτό σε αλληλεγγύη με κάποιους παραγωγών ε, καθώς και των διαφόρων φορέων στον τομέα του τοπικού γάλακτος. Και βεβαίως να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις που είναι προς όφελος των τοπικών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποφύγουμε τις ε, αρνητικές επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια, οικονομική αυτονομία ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων. Το σλόγγαν μας σήμερα είναι ότι το τοπικό γάλα... Κύριο Τσούτερ είναι αντιπρόεδρος μιας οργάνωσης στο περιβάλλον, ε, τη χρήση και την κατανάλωση κρέατος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα σας δώσω μια εικόνα που είναι πιο ευρεία και πιο πολιτική από αυτήν που μας παρουσίασε η καθηγήτρια περίπτωση Θα ξεκινήσω θυμίζοντάς σας ότι η ΚΑΠ είναι πολύ δύσκολο να εξολογηθεί σε ένα πλαίσιο σαν και αυτό, γιατί το να για να αξιολογήσουμε τις ε, επιπτώσεις τη αναπτυσσόμενες χώρε πρέπει να συγκρίνουμε που έχει αυτό ο αντίκτυπο στι διάφορε χώρε όσον αφορά τη χρήση τη γη των υδάτων. Είναι, επομένως, είναι, πολύ, είναι πολύ δύσκολη η εργασία. Θα σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε η ΚΑΠ το 1961, η την ηγεσία του Μάντσχολτ, ο κόσμος ήταν διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Σας δείχνει τη δημογραφική εξέλιξη μεταξύ του 1900 και 2020 και βλέπουμε και τι περιμένουμε για το μέλλον. Και όταν ξεκίνησε η ΚΑΠ, είχαμε μια ραγδαία ανάπτυξη του πληθυσμού. Άρα χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγή, να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, ταΐσουμε αυτό την την, να καλύψουμε αυτή την μεγάλη ανάγκη. Βλέπετε λοιπόν από τις ευκαιρίες που τους παρέχει το εμπόριο. 300 εκατομμύρια είναι φτωχοί των πόλεων. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό που βασίζονται σε μικρές παραγωγικές μονάδες και που πουλάνε σε τοπικές αγορές, γιατί οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν στις προσπάθειες εξαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλη. Όχι μόνο τα νομιστικά εμπόδια, αλλά και η διάσταση της κλίμακας που δεν μπορούν να πετύχουν για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί στις αγορές και για να ε, δείξουν ενδιαφέρον μεγάλοι αγοραστές. Ωστόσο, στον κόσμο σήμερα οργανισμού γεωργίας, οι πιο πολλές παραγωγές έχουν να κάνουν και προορίζονται για εξαγωγές για κάποιες καλλιέργειες αυτό είναι πολύ εξωσμίωτο, όπως είναι για τα φασολία της σόγιας. Έχουμε εκατομμύρια τόνων κοινωνικής παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγές. Είναι επίσης πολύ σημαντικά τα ποσοστά αυτά και για τη ζάχαρη, το φινικέλαιο και για άλλα προϊόντα που βλέπετε στο γράφημα. Αυτές οι εξαγωγές δεν γίνονται από μικρούς καλλιεργητές που άλλους ε, παίκτες του παγκόσμιου εμπορίου και που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες εξαγωγών. Ισπλοκο θέμα και από τις δύο πλευρές ε, του διαλόγου υπάρχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Το εμπόριο ενθαρρύνει ε, τις χώρες να εξειδικεύονται σε αυτό που είναι καλύτερο για αυτές ως προς την παραγωγή. Πολλές φορές εκεί υπάρχει και αγοραστική δύναμη. Συχνά βλέπουμε ε, φτωχέ χώρες που έχουν ε, επιστηστικό έλλειμμα και παρόλα αυτά εξάγουν γιατί αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τους εξαγωγείς. Επίνω περισσότερες εισαγωγές. Θα πρέπει να αποκεντρωθεί λοιπόν, υπάρχει το επιχείρημα ότι πρέπει να αποκεντρωθεί παραγωγή για να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ αυτέ τι περιοχέ. Ε, όσον αφορά τη συνεργασία μου τώρα με τον ΟΗΕ και τα συμπεράσματα που έχω, βλέπετε, έχουμε τις εξαγωγέ από τη μία και από την άλλη την παραγωγή για την ε, κάλυψη των τοπικών αναγκών. οι μικροί παραγωγοί δεν τα καταφέρουν και αναγκάζονται να αυτό το φαινόμενο. Το 90 λοιπόν και το 2000 το 2000 χρειάστηκε να γίνουν τις αγωγές τροφίμων και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι αυξημένες αγωγές δημιούργησαν μεγάλη εξάρτηση από τις αγωγές για να εξασφαλιστεί Λοιπόν, πως πληθυσμοί σε πολλέ αντισόμενες χώρε, ειδικά στην Ποσαχάρη Αφρική και σε κάποια σημεία τη Νότια Αφρική, έχουν ε, εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγέ για την κάλυψη των αναγκών του. Η Αφρική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί παρά τον μεγάλο οι εισαγωγέ έχουν αυξηθεί γιατί η, ανα... η πληθυσμού ήταν πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί να υποφερθούν από αυτό βραχυπρόθεσμα η φτωχή των πόλων, αλλά μακραπρόθεσμα όμως των εξαγωγών. Η γεωργική παραγωγή που προορίζεται στην εξαγωγή είναι βιοχρονοποιημένη και δημιουργεί ε, προβλήματα περιβαλλοντικά όπως είναι η διάβρωση, την ε, ε, Επίσης το έδαφος δεν είναι τόσο γόνιμο για καλλιέργειες και έτσι πάλι δημιουργείται, συνεχίζεται αυτός ο κύκλος για την ανάγκη εισαγωγών και επίσης χρειάζονται, χρειάζεται και η χρήση παραστοκτώνων. Βλέπεις 14 30 χρόνια χωρίς του χάρτη. Βλέπουμε σε αυτό το χάρτη την αύξηση της παχυσαρκίας. Αυτή είναι μια αξιολόγηση που βασίζεται στους πληθυσμούς 20 χώρων. 90 Νότια Αφρική η παχυσαρκία έχει αυξηθεί. 800 εκατομμυρία είναι υπέρβαροι. Και αυτό αφορά το 2,8 του παγκόσμιου ΑΕΠ. Γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί τα γεωργικά προϊόντα που ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις είναι προϊόντα τα οποία είναι επεξεργασμένα. Η βιομηχανοποίηση λοιπόν των συστημάτων ε, επισήτησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που ε, επηρεάζουν αρνητικά τους βυτικούς πόρους ε, των κατοίκων στις αναπτυσσόμενες το παράγουν πολύ περισσότερο ένα εκτάριο ανά άτομο και χωρίς με εξαγωγικές επιδοτήσεις είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στην παραγωγή κρέατος, ε, γάλακτος κτλ. όπως στην Μπουρκίνα Φάσο παραδείγματος χάρη και θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να δούμε ποιο ε, εποφελείται, ποιος χάνει από το αυξημένο εμπόριο. Να δούμε ποιοι είναι οι λιγότερο ανταγωνιστικοί. Ε, αυτές οι χώρες εισάγουν από εμάς. Και όσο περισσότερο το κάνουν αυτό, τόσο λιγότερο θα έχουν το κίνητρο ε, να επενδύσουν ε, για την ε, ανανέωση των τοπικών συστημάτων επισήτηση. Θα πρέπει να σε λιγότερη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και βοηθάνε στην μείωση της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους και για τους πανελίστες και για την κυρία Πλάνκο, η οποία πήρε το λόγο Μαρία, μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Ε, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο στην έρευνα και στα αριθμητικά στοιχεία που σας έδωσα. Βλέπετε την τιμή των ε, εισαγωγών και των εξαγωγών. Όχι ποιος ωφελείται. Στην έρευνα θα δείτε πιο πολλές ε, λεπτομέρειες και ένα τομέα όπου αναλύουμε και σχολιάζουμε έρευνες που ακριβώς αναλύουν πώς εξέλιξε το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και πώς υπάρχει και αρνητικός αντίκτυπος. Το σχολίασα, αλλά εντάχει Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι χώρες ε, επικεντρώνονται σε προϊόντα εξαγωγής. Ε, αυτό έχει αρνητικέ επιπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις για τον τοπικό γεωργικό πληθυσμό και για την παραγωγή. Έχετε δίκιο. Και αυτό έληφθη υπόψη στην έρευνα. Επίσης, Το θέμα είναι αυτό συμβαίνει λόγω της κοινή πολιτικής. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται λόγω της ΚΑΠ ή του τοπικού θεσμικού πλαισίου προφανώς στις χώρες αυτές. Τι ευθύνη φέρει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Ο κύριος Νόιχλ. Θα ήθελα... Ο κύριος Νόιζερ, συγγνώμη να ευχαριστήσω τους ε, τρεις ε, πανελίστες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάθαμε στοιχεία πολλά, γιατί αυτή η κοινή συνεδρίαση μας καταδεικνύει ότι όλο και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη στην υποσαχαρή Αφρική. Χάρηκαμε δηλαδή σε μικρά προγράμματα προγράμματα τα οποία ωφελούν ε, τις γυναίκες. Παρόλα αυτά, αναγνώσει σε ό,τι αφορά, ε, για παράδειγμα, και τα θέματα αναγκών ε, σε σκόνη γάλακτος, γιατί είναι τεράστια και τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τις τρεις παρουσιάσεις. Εγώ θα ήθελα Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό που λαμβάνει η χώρα σήμερα αυτή η συζήτηση, όπως γνωρίζουμε και θα ξέρετε κι εσείς. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ε, συζήτησης ε, για την ε, μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής και στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γεωργίας, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν σε άλλες συζητήσεις, συνεχώς μας λένε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αναφέρεται ότι η Ευρώπη θα πρέπει με αυτό που συζητάμε και ακούμε εδώ, σε ό,τι φορά τον αντίκτυπο δηλαδή. Δεύτερον, ε, είναι στα πλαίσια της κοινή δικής πολιτικής της υπάρχουσας, μεταφέροντας τις ενισχύσεις από τη μία πλευρά στην άλλη, ή υπάρχουν άλλες λύσεις, διότι εγώ θεωρώ ότι να αλλάξουμε στο βορρά και στο νότο, έχουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως η γεωργία ε, των μικρών παραγωγών ξαφανίζεται σιγά σιγά και στην Ευρωπαϊκή γιατί μια μελέτη όπως η δική σας ε, δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο, δεν αναφέρει τίποτα εκτός του πλαισίου της υπάρχουσας κοινή γεωργικής. Υπάρχει ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε στο πρώτο ερώτημα. Η κυρία Μπλάνκο θέλει να απαντήσει το δεύτερο. Έγινε ένα ερώτημα προηγουμένως. Θέλετε να απαντήσετε. Αφορούσε το σύνολο του πάνελ. Ναι, φαντάζομαι θα έχουν και συνάδελφοι να πούν πολλά. Η αντίδρασή μου πάντως αφορά και το τελευταίο ερώτημα. Ε, εγώ θεωρώ ότι η προτεραιότητα σήμερα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να θρέψει τον κόσμο, αλλά να συνεισφέρει ε, έτσι ώστε η κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια να μπορεί να θρέψει τον εαυτό της. Όχι να πάνε προς την αυτάρκεια, έτσι. Δεν είναι αυτό επιθυμητό, δεν είναι καν πραγματοποιήσιμο. Αλλά να μειωθεί η εξάρτητη τοπική οικονομία η δημιουργία αυτών των δυνατοτήτων μέσω της ε, επανικοδόμησης τοπικών συστημάτων διατροφής είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όμως πολλές αναπτυσσόμενες χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πολιετές σχέδιο έτσι ώστε, όχι, ώστε να μην είμαστε πάντα όμοιροι ε, του βραχυπρόθεσμου και να λέμε ότι θα την παγκόσμια. Ε, ναι, κυρία Μπλάνκο, παρακαλώ. Ναι, έφερε κάποια αποτελέσματα της μελέτης ότι αν αυξηθεί δηλαδή η παραγωγή αυτή τη στιγμή, ε, τότε θα μειωθούν παγκοσμίω. Ε, για να έρθω τώρα... Ε, εντάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι για να γίνει αυτό, αλλά δεν ήταν ο στόχος της μελέτης να βρεθούν άλλοι τρόποι. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικό, το οποίο ανέφερα και στις συστάσεις ε, χρειαζόμαστε μια πιο συστηματική προσέγγιση ότι αφορά τι πολιτικές μας. Αυτό δεν αφορά μόνο τη γεωργική πολιτική, διότι είναι η γεωργική πολιτική οι πολιτέτες τη συστάσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό, αυτό τον αντίκτυπο ε, τον διατομεακό, ε, διότι υπάρχει ασυνέπεια αυτή τη στιγμή. Ε, θέλουμε να προωθήσουμε το εισόδημα των γεωργών, και να εξετάζουμε μόνο αυτό και αυτόν τον στόχο, δεν βλέπουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Παραδείγματο. Γνωρίζω βεβαίω ότι δεν είναι αυτή η λύση που εσεί περιμένατε, αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά αλλάξουμε την προσέγγιση μα, εάν αρχίσουμε να εξετάζουμε τη γεωργική πολιτική από κοινού με άλλε πολιτικέ, την πολιτική ενέργεια, την πολιτική εμπορίου, την εμπορική πολιτική, την πολιτική ανάπτυξη και είναι δύσκολο βέβαια αυτό να δούμε όλε. Ήταν εξαιρετικά συμπληρωματικοί στι παρεμβάσει του και δείχνουν το εξή. Ε, το ερώτημα που θα θέσω μάλλον στην κυρία Μπλάνκο πρώτα, διότι είναι και οικονομολόγο και ασχολείται με τα γεωργικά, τι κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια. Εγκαταλείπουμε του μηχανισμού ρύθμιση τη αγορά. Εγκαταλείψαμε τι ποσοστώσει. Τι συμβαίνει σήμερα με το γάλα, παραδείγματο χάρη, που δεν υπάρχουν, υπάρχουν ποσοστώσει. Έχουμε υπερπαραγωγή. Και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για τους ε, γεωργούς, οι οποίοι γίνονται πιο φτωχοί. Τι συμβαίνει στην Αφρική. Ο κύριος τα είπε πολύ σωστά και τα ξέρει και ο Λιβέντε Σιούτερ αυτά πολύ καλά. Ήταν και εισηγητή στα Ηνωμένα Έθνη για ζητήματα διατροφή. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Αφρική. Του εξάγουμε εμεί γάλα σε σκόνη, διότι ψάχνουμε αγορέ, αφού έχουμε ε, πλημμυρίσει από γάλα σε σκόνη και εκεί έτσι φτωχοποιούνται οι Γεωργοί οι Αφρικανοί που θα μπορούσαν εκεί. Οι Καναδοί ήταν πολύ ευφύ, δεν δέχτηκαν να ανοίξουν την αγορά γάλακτο. Είναι κλειστή. Έμεινε κλειστή η αγορά γάλακτο και εμεί θα του εξάγουμε ε, καμαμπέρ στα, στην ακτή τη Δυτική Αφρική, Λακτάλη, Νεστλέ, Ντανόν, Αρλά. Βλέπουμε εδώ όλα τα μεγαθύρια. Τι συμβαίνει λοιπόν, εντάξει, όσο γίνεται μεγαλύτερη αυτάρκεια στον κόσμο, αλλά κυρίω να έχουμε μηχανισμού ρυθμιστικού σε ό,τι αφορά τι τιμέ. Δεν μπορεί να, μιλάμε, να λέμε καν τη λέξη ποσόστοση, διότι. Ε, η Μαρία. Ε, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Η κυρία που μίλησε πρώτη είπε ότι αξιολογείται τώρα τι πολιτικέ που εφαρμόζονται. Με ενδιαφέρουν με ενδιαφέρει πώ εξηγείται τα παλιότερα συστήματα. Τώρα δεν έχουμε εξαγωγικέ επιδοτήσει, να το γνωρίζω, αλλά από το 2009, από το που καταργήθηκαν οι επιδοτήσει ε, για το κοντόπολο, η αγορά στην Αφρική τετραπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξουμε την πολιτική μας είναι ένα σύστημα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει και το οποίο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Η δική μας η αγορά, καθώς και η Αμερικάνικη αγορά, έχουν ενισχυθεί γιατί υπάρχει μια πολιτική αποκλεισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ τα έχουν και αυτές το δικαίωμα να κλείσουν τις δικές τους αγορές. Δεν έχει όμως να κάνει με το να τους βοηθήσουμε, αλλά να τους βοηθήσουμε συστηματικά. Ευχαριστώ. Δασμού στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτό είναι θέμα τη Μπουρκίνα Φάσο. Αν θέλει να υπάρχουν μηχανισμοί για να επιβληθούν τα ζωσιμότητα των δικών μα συστημάτων. Και το είπαν και οι άλλοι Ιρλανδοί συναδελφοί. Εξαγάγουμε. Ευχαριστώ κύριε Μιούλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μιούλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν ε, έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να καταργήσουν ε, τις ενισχύσει αυτές και σε ό,τι αφορά τις πρωτεϊνούχες καλλιεργίες. Ζήτησα να μου φέρουν τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία. Όντως έχουμε πριν να έχουμε μείον το πώς μπορούμε να ασκήσουμε βιώσιμη πολιτική και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις τοπικές οικονομίες. Να... Αυτό το θέμα μας απασχολεί πολύ, να υποστηρίξουμε και στις γαλακτώσεις σκόνη. Κύριε Σκούτερ, είπατε ότι θα θέλετε να υπάρχει ένας μηχανισμός προειδοποίησης. Uh, uh, ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι ε, σε κάποια κράτη-μέλη που εξαρτώνται άμεσα από αυτή τη μορφή ενίσχυση. Ε, στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη, υπάρχει αυτή η ενίσχυση για το χείριο κρέα, για, για τα πουλερικά και αν δεν υπήρχε, ο συγκεκριμένο κλάδο δεν θα ήταν βιώσιμο. Έχετε ε, την ε, ευρωπαϊκή αγορά και με αρνητικό τρόπο. Γιατί το λέω αυτό. Η παραγωγή των χωρών Μερκοσούρ δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες απαιτήσει, τις ίδιες προδιαγραφές ε, για ένα κιλό κρέας σε σχέση με τις δικές μας προδιαγραφές στην Ευρώπη και αυτό παράγεται με πάνω από 3 ευρώ. Είναι λοιπόν σημαντικό να δημιουργήσουμε τοπικές δυνατότητες παραγωγής. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή εισάγει τρόφιμα αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι εξαγωγές μας είναι μόλις 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αλήθεια ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιδράσουν. Ολοσμένες φορέ, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να, να σταθούν απέναντι σε έναν ανταγωνισμό ο οποίο καταστρέφει ολόκληρου τομεί. Κύριο Ντέ, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ για τι παρεμβάσει. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω προ τον κύριο Ντιάλο, Καταρχά, πρώτη ερώτηση. Μιλήσατε για τη σκόνη γάλακτος που εμπλουτίζεται και είπατε ότι αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Μπορείτε να επιδράσετε, να επηρεάσετε την κυβέρνησή της προκειμένου. Ποια εμπόδια, τι ρυθμιστικά εμπόδια υπάρχουν, μπορείτε να μας πείτε. Τρίτη ερώτηση. Θα σας ωφελούσε αν με την αναπτυξιακή βοήθεια για τις επενδύσεις ε, στις μικρές γαλακτοκομικές αυτές επιχειρήσεις ε, μπορούσαμε να πετύχουμε μία ενίσχυση για να πρώην ε, πρόεδρο της ε, Σχετικής Επιτροπής από το Πανεπιστήμιο του Χάμπελ της Γερμανίας. Αλλά... Καλώς ορίζουμε τον κύριο Χαραντφον Βίτσε. Το πολύ. Εκτός μικροφώνου, κύριο κύριος Βίτσε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση Ο στόχο του άρθρου 28 τη Συνθήκης της Λισαβόνα έχει στόχο τη μείωση και την εξάλληψη της φτώχειας. Η φτώχεια, η πείνα σχετίζονται γιατί οι περισσότεροι υποσυντισμένοι ζουν στην Ήπεθρο είναι ιδιοκτήτες μικρή, μικρών εκτάσεων δεν έχουν, ή δεν έχουν γη. Και η γεωργία είναι το κλειδί για την μείωση της πείνας και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχω διδάξει οικονομική ανάπτυξη για πάνω από 30 χρόνια και έχω 60 ώρες σημειώσεων και διαλέξεων, αλλά θέλω να συνοψίσω λίγο αυτές τις 60 ώρες σε δύο προτάσεις. Μακροπρόθεσμα, η κινητήριος δύναμη της αγροτικής ανάπτυξης και για τη μείωση της πείνας στον κόσμο είναι η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε γνώση και σε δεξιότητες. Και το δεύτερο είναι χρηστή διακυβέρνηση, λειτουργική οικονομία της αγοράς και τα κατάλληλα διεθνή συστήματα. Επίσης ανακαλύψαμε ότι η φτώχεια και η πείνα είναι έντονες στις περιοχές όπου οι αγρότες έχουν ε, ελλειπή πρόσβαση σε τεχνολογίες που πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια. Όπως είναι τα λοιπάσματα. Θα εστιάσω λοιπόν το θέμα των τιμών της κίνησης της αγγελικής πολιτικής. Και θα ξεκινήσω μια παρατήρηση. ότι η μείωση των τιμών σημαίνει και μία αλλαγή που δείχνει ότι το 2000 οι τιμές έχουν αρχίσει να αυξάνονται και ο λίγος είναι ότι σε παγκόσμια κλίμακα η ζήτηση ξεπέρασε σε ρυθμό την ανάπτυξη της προμήθειας. Υπάρχει μεγάλο κενό εισαγωγών σε πάρα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι χώρες περνάνε μια φάση οικονομικής ανάπτυξης που πέρασε η Αγγλία την εποχή του Ρικάρντο όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπερνάει την ε, ικανότητα απορρόφησης από την αγορά. Αυτές οι εξελίξεις στην αγορά που ανέφερα δημιουργούν πολλές ανησυχίες για την επιστημική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και το κόστος είναι πείνα, πολιτική αστάθεια, μετανάστευση και βία. Η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται ραγδαία και θα πρέπει να καλύψουμε αυτή την ζήτηση για προϊόντα αγροτικά, επεκτείνοντας τη γη ή παράγοντας περισσότερα στην γη που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Η επέκταση των εκταριών δεν είναι εφικτή γιατί είναι περιορισμένη η γη σε παγκόσμιο πεδίο. Οι πιο παραγωγικές γης ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλά τμήματα του κόσμου. Δεν υπάρχουν αποθέματα ε, γεών για τη γεωργία. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, περιοχές όπως είναι το τροπικό δάσος για τέτοια χρήση. Αύξηση τη παραγωγή για την κάλυψη των αναγκών θα πρέπει να προέρχεται κυρίω από την απόδοση. Ο ΦΑΟ ε, αναμένει 9% ε, αύξηση από την απόδοση περισσότερο και όχι από την επέκταση της χρήσης της γης. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας έχει μειωθεί από την Πράσινη Επανάσταση Μπόρλο το 1960 και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Θα αναφέρω τρεις λόγους που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ένας είναι ότι παρμελούμε την γεωργική έρευνα η έρευνα αυτή ξεκίνησε στα τέλη τη δεκαετία του 90 όταν άρχισαν να σωρεύονται τα πλεονάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερο λόγο είναι, είναι ευξενόμενοι περιορισμοί στη χρήση τεχνολογιών όπως είναι η παραδοσιακή η γενετική τεχνολογία ή η προστασία των καλλιεργιών. Και τέλος έχουμε πολύ πετυχημένο λόμπινγκ από συγκεκριμένε ομάδες οι οποίες προτιμούν την χαμηλή παραγωγικότητα. Το αυξανόμενο εισαγωγικό κοινό των φτωχών χωρών θα μπορούσε να κλείσει μόνο αν οι πλούσιες χώρες παράγουν περισσότερο και εξάγουν περισσότερο φαγητό. Και όχι λιγότερο, όπω λένε κάποιοι, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά θα ήταν τα ωφέλη αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματούσε να είναι ένας ο μοναδικός καθαρός εισαγωγές προϊόντων. και να αξιοποιήσουμε την δική μας βιομηχανία τροφιμών. Αυτές τις εισρωές αγροτικών προϊόντων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Βλέπετε λοιπόν, μεταξύ 17 και 34 εκατομμυρίων εκταρίων είναι το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της χρήσης με στον υπόλοιπο κόσμο. Ας προχωρήσουμε στις επιλογές. Είναι προφανής και είναι ότι η ερευνητική πολιτική στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Αυτά τα πρέπει να είναι ε, κοινό στοιχείο της, ε, κεντρικό στοιχείο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα ωφέλη για την κοινωνία είναι πολύ υψηλά, όπως βλέπουμε προς το παρόν, σε οικονομικούς όρους. Υπάρχουν θετικές εξωτερικότητας, οι οποίες υλοποιούνται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και δικαιολογούν φυσικά την ε, χρηματοδότηση ερευνών. Μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα μια επιδότηση πιγκού, όπως ε, την ονομάζουμε με οικονομικούς όρους. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη ξεπερνούν ε, τις επιπτώσεις στην κοινωνική πρόνοια. κάθε ποσοστό απόδοση θα είναι υπέρ της ε, κοινωνίας. Θα αυξήσει την ε, κοινωνική πρόνοια κατά 500 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ωφελεί και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, αλλά θα μειώσει την εισαγωγή εικονικής αγροτικής αρρώσιμης γης κατά 1,2 εκατομμύρια εκτάρια. Επίσης αυτό θα διατηρήσει 1,2 εκατομμύρια εκτάρια φυσικών ενδιατημάτων. Θα μειώσει τις εκπομπές του του άνθρακα κατά 220 εκατομμύρια τόνους. Και αυτό φυσικά υποφελεί σε μεγάλο ποσοστό την κοινωνία ε, σε βαθμό 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό θα, δημιουργήσει στην, θα βοηθήσει τη δημιουργία 600.000 εκταρίων τροπικού δάσους. Όσον αφορά την ψυχική ασφάλεια και την φτώχεια στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, πολλές φορές ακούω το επιχείρημα Πώ το υπολογίζετε ότι αυτό έχει γίνει έτσι, αν εμεί ξεκινήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγουμε περισσότερα, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την απόδοση και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε και την εντατικοποίηση της ε, καλλιέργειας. Και η απάντησή μου είναι ότι η εντατικοποίηση της χρήσης της γης δεν θα πρέπει να είναι ούτε καλή, δεν ούτε καλή κακή, πρέπει να είναι βιώσιμη. Λοιπόν, το μελετήσαμε αυτό το θέμα και είδαμε ότι η τη απόδοση για συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι ίδια. Ας δούμε λοιπόν στο σιτάρι, στη στηρά. Κατά τη διάρκεια της ε, έρευνάς μας από το 2003 στο 2013 υπήρχε μια ανάπτυξη ετήσια στην απόδοση κατά 0,86% και αυτή θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα πιο δικοπημένη παραγωγή, με περισσότερα λοιπάσματα κτλ. Ή θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα καινοτομία και την κοινοτομία την μετράμε με την αλλαγή του TFP, Total Factor Productivity, που μετρούν την ε, παραγωγή και βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση της απόδοσης ε, συνδυάζεται με μειωμένη εντατικοποίηση της χρήσης της γης. Άρα το συμπέρασμά μου και η σύστασή μου είναι να μην ασχοληθούμε πλέον με την ιδέα της βιώσιμης εντατικοποίησης, γιατί το αντίθετο ακριβώ ισχύει. Είναι ε, ένα, μέτρο που ακολουθήθηκε από άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες ε, Πολιτείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι βλέπουμε την οικολογική γεωργία που θα μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα ε, πολιτική γιατί το μισό της σύγχρονης καλλιέργειας ε, ε, είναι τέτοιου τύπου καλλιέργεια, οικολογική καλλιέργεια. Αυτό σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει η συνολική αρρώσμη γη να επεκταθεί κατά 70 εκατομμύριο εκτάρια με μεγάλο κόστος για την κοινωνία, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες περιοχές, απώλεια ενδυτεμάτων, βιοπικιλότητας και άλλες συνέπειες που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή. Παρατήρησα ότι κάποιοι συναδελφοί είχαν πάνω από 10 λεπτά. Θέλετε να σταματήσω στα 10 λεπτά. Επιτρέψτε μου κύριε Βίνκε, παρακαλώ να τελειώνετε και κύριε Μαρ, αφήστε τον να τελειώσει. Συχνά ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν να ακούμε, αλλά πρέπει να μπορούν να μιλήσουν όλοι. Τελειώνετε παρακαλώ. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη... Λοιπόν, είναι κακό για τους ε, φτωχού και τους πεινασμένους, Γιατί η μειωμένη παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήνει τι τιμέ των γεωργικών προϊόντων. Περισσότερο από ποτέ η κοινή αγροτική πολιτική και αποφάσει ειδικέ θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις και όχι σε ομάδες ε, άσκησης πίεσης. Θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να καταστήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και πάλι αξιόπιστη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Βίκε. Και τώρα θα πρέπει να περάσουμε αμέσως, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα περάσουμε αμέσως λοιπόν στο επόμενο πάνελ που είναι τα συμπεράσματα ε, της σημερινής συζήτησης είναι και ο Επίτροπος Χόγκαν εδώ. Τα συμπεράσματα λοιπόν για την ε, ε, συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη. Λοιπόν, για να μην χαθεί χρόνος και να μπορέσουν να παρέμβουν έστω και για λίγο οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο αμέσως στον Επίτροπο, στον κύριο Χόγκαν, να μας κάνει την παρουσίασή του, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμοι ε, καλεσμένοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ. Χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα. Η κατανόηση ότι αποτελούμε μέρο ενό παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Γνωρίζουμε τι προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Ε, η κοινή γεωργική πολιτική ε, ε, Ευρωπαίου γεωργούς. Ε, δεν συμβαίνει όμω αυτό πια. Είναι παρελθόν η πολιτική μας η γεωργική συνδέεται και ευθυγραμμίζεται με, τις, με, τις, με τους στόχους της ανάπτυξης. Υπάρχουν ακόμα κάποιες ενισχύσεις. Θα έρθουμε, θα έρθουμε σε αυτό. Πολύ κάτω από την τιμή παραγωγής. Ε, και λαμβάνουμε υπόψη τις παγκόσμιες τιμές. Οι εξαγωγικές επιστροφές δεν υπάρχουν πια. Την 1η Νοαρίου του 2014. Να έχουμε κανόνες ε, ίσους για όλους στο εμπόριο. Έχουμε πολύ καλές ε, ε συνθήκες πρόσβασης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, αδασμολόγητες ε, για τις, λιγότερο, για τις πιο φτωχές χώρες ε, και μονομερείς συμβάσεις με τις φτωχές χώρες. Έχουμε εμπορικέ συμφωνίες έτσι ώστε να μπορούν οι πιο φτωχές χώρες να προστατεύουν τις ευαίσθητες παραγωγές τους. Υπάρχουν παγκόσμιες δικλείδες ασφαλείας για να μπορούν να υπερασπίζονται και να αμήνονται απέναντι στι εισαγωγέ. Είπε ένα ομιλητή σήμερα ότι μπορεί να φάσω κάποια πράγματα ε, να πω ότι στα πλαίσια των οικονομικών, των οικονομικών συμπράξεων και σχετικών ε, συμφωνιών Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα έλεγα να το κάνετε έτσι ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε αυτέ τι ευκαιρίε εφόσον το επιθυμείτε. Παραδείγματο χάρη, η κυβέρνηση να φάσει θα μπορούσε να θέσει ένα δασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει την απόφαση που πρέπει να πάρθει από μια κυριαρχική κυβέρνηση. Επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει μονομερώς ε, Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ιαπωνία μαζί. Έχουμε λοιπόν συνεργασία μεταξύ ε, γεωρικής πολιτικής, πολιτικής ανάπτυξης και συμπαίκτε μα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Στην ανακοίνωσή μας ε, του Νοεμβρίου υπάρχουν πολλές σκέψει για το πώ μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε περισσότερα με την κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει σε δέσμευση ε, μια για μια ισορροπημένη εμπορική πολιτική. Η, η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο για να επιτευχθούν ε, οι στόχοι τη ε, σύνο κορυφή τη Βαλέτα μεταξύ με αυτέ τι μη, μη τακτικέ και μη ελεγχόμενε ροέ μετανάστευση. Να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τι προκλήσει που έχουν να κάνουν με την παράτυπη μετανάστευση σε οικονομικό επίπεδο, να μείνουν οι νέοι άνθρωποι εκεί. Έχω ήδη αναφέρει τον θετικό αντίκτυπο των εξαιρετικά ευνοϊκών ε, Μια ευκαιρία στα πλαίσια του προγράμματος εξωτερικών επενδύσεων ε, για, τις, ε, για τον αγροτικό τομέα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ύπεθρος είναι πολύ σημαντική για την γεωρική ανάπτυξη, για την οικονομική, αυτό το αυξανόμενο εργατικό δυναμικό. Αυτό θα αυξήσει και την προσφορά, θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητα της αφρικανικής γεωργίας με υποστήριξη και για τα μικρά γαλακά με το στηρό, με το 2016. Υπάρχουν τα μοντέλα παραδοσιακής συνεργασίας για την ανάπτυξη ε, και τώρα επικεντρωνόμαστε στο να εστιάσουμε στην... Είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να είναι μια πραγματική ευκαιρία η Γεωργία για τους νέους στην Αφρική. Η, η, όλα αυτά, όλες, αυτές τις εκδηλώσεις που οργανώσαμε ε, και με τον Επίτροπο εμεί ζητήσαμε από τους γενικούς διευθυντές ε, από κοινού να ετοιμάσουν μια task force για να προκύψουν συστάσει και προτεραιότητε για τα επόμενα βήματα στην γεωρική συνεργασία με την αφρικη συνολικα Ώστε 10-11 πυρογνώμονες να συνέλθουν από κοινού και να έχουν τακτικέ συνεδριάσει και ω το τέλο του έτου να μα παρουσιάσουν μια έκθεση. Θέλω πραγματικά να το κάνουν αυτό σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να αναφέρω ότι ξεκίνησε ήδη ο διαγωνισμό ε, για την προκήρυξη των θέσεων. Πως ε, παρουσίασε καλά τα πράγματα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε μια, ένα καλό ιστορικό για την Αφρικανική, για την ε, αναπτυξιακή, ε, την ανάπτυξη στην Αφρική. Ακούμε σήμερα το απόγευμα πολλά για τον πολιτικό χώρο, για την ανάγκη ρύθμισης, ε, για τα μέσα και τα μέτρα αποζημίωσης Ελπίζω να κατέστη σαφές ότι ακόμα και στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης που έχουν δημιουργήσει μεγάλο φόβο στον τομέα παραγωγή τροφίμων και τον αγροτικό κλάδο, υπάρχει σαφής ε, περιθώριο για τις χώρες να σχεδιάσουν τις πολιτικές τους και τις στρατηγικές τους μετρέπω τον κλάδο σε όλες τις τα επίπεδα, τον αγροτικό κλάδο και τον ε, κλάδο των τροφίμων. Έχουμε 9 δις ευρώ για την περίοδο αυτή. Υπάρχει σαφής ε, δημοσιονομική υποστήριξη, ιδιαίτερα στη Αφρική, για να υποστηριχθούν οι τομεακέ ενισχύσει με το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων. Επιτυχικό κλάδο έχει δυνατότητα να δυναμητήσει την τομέα αυτών, ο οποίος, όπως είπε ο Επιτροπός, έχει μείνει σε χαμηλά ποσοστά επενδύσεων. Χρειαζόμαστε πολλούς ε, επενδυτές ε, και υπάρχει επένδυση, ξέρετε, στην ψηφιακή εποχή και σε πολλούς άλλους κλάδους, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, όχι όμως τόσο πολύ στα γεωργικά. Γι' αυτό λοιπόν σκοπός είναι να προσπαθήσουμε να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα, να υποστηρίξουμε τους ντόπιου νεαρούς επιχειρηματίες προκειμένου και με την γραμματεία και με τον iPad, το για να εντοπίσουμε τους κλάδους εκείνους και τις οικονομικές δραστηριότητες, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εντό του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, προκειμένου να τους χορηγήσουμε υποστήριξη. Υπάρχει ένα μεγάλο δυσί. σε επαγγελματικού όρου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε τους όρους πλαίσιο. Αναφέρατε, ε, κύριε καθηγήτα, την αγροτική έρευνα. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε από ότι σε ό,τι αφορά τις... Ε, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις όπου θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε διάφορους τρόπους για να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στους κλάδους αυτούς, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και στη διατροφή. Όπως ξέρετε,